Μπορούμε να ψηφίσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η πρώτη έκθεση είναι η έκθεση Ριμπέιρο. Ονομαστική ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι. Cred că acum a votat toată Ψηφίσατε όλοι. τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Συνεχίζουμε. Γκάρδια Ζαμπάλ Ρουμπιάλ. Είναι η επόμενη έκθεση που ψηφίζουμε. Και πάλι ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ.